Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει τι απαραίτητε μεταρρυθμίσει και μόνο τότε μπορεί να αποφασίσει αν θέλει να παραμείνει ανεξάρτητη και αυτόνομη ή να ενσωματωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ κύριε Μέλτσερ. <clears throat> Ακολουθούν οι υπόλοιποι ομιλητέ. Καταρχήν ο κύριο Γκάλερ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. <clears throat> Πράγματι υπάρχει